Thank Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κάποτε είχα την ιδέα ότι μπορούσα να γίνω ευρωβουλευτής, αλλά εδώ δεν μπορώ να ανάψω τα μικρόφωνα. Ε, καλύτερα είμαι πρόεδρος της ΕΤΕΠ, διοικητής της ΕΤΕΠ. Ευχαριστώ. Ήρθα να σας μιλήσω για το θέμα της, του πρασινίσματος της ΕΤΕΠ ε, και ε, πριν από την COP21, ε, 25 συγγνώμη, φαίνεται πως πάντοτε Μπορούμε να επηρεάσουμε τις ε, συζητήσεις στην ΚΟΠ και ελπίζω πως το ίδιο θα συμβεί και φέτος. Ε, είμαι ευγνώμων ε, στον ε, κύριο Καμφάν που μου δίνει την ευκαιρία σήμερα να σας μιλήσω. Την περασμένη εβδομάδα εσείς υιοθετήσατε ένα ψήφισμα που δήλωσε ότι το θέμα του κλίματος είναι έκτακτης, είναι μάλλον κατεπήγον, συμφωνώ μαζί σας και πιστεύω πως πρέπει να εκμεταλλευτούμε το τελευταίο παράθυρο ευκαιρίας πριν από καταστροφικές κλιματικές αλλαγές. Αυτό αληθεύει και το αναφέρω για την προστασία και των, οικοσυστήμα, των οικοσυστημάτων και της βιοπικιλότητας, διότι έτσι θα δημιουργηθεί ένα ε, βάθρο για την ε, κατάσταση που πριν τον Οκτώβριο του 2020 ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, κλιματικές αλλαγές και την κρίση του κλίματος αλλά μπορούμε πιστεύω να το αντιμετωπίσουμε αυτό αρκεί να ενεργήσουμε οργανωμένα και συντονισμένα. Είχαμε μία εξέλιξη στην ε, τράπεζα που εξέπληξε τους πάντες ε, συμπεριλαμβανομένων και ημών που είμαστε στην ε, διοίκηση της τράπεζας γιατί γνωρίζαμε πως ήταν δύσκολο το πράγμα όταν 28 κράτη-μέλη δεν έχουν βέβαια πάντοτε ε, τις ίδιες ιδέες και την σύγκληση που είναι απαραίτητη ειδικά για τέτοια δύσκολα ζητήματα όπως αυτό τελικά όμως καταφέραμε να αποσπάσουμε τεράστια πλειοψηφία και από τους ε, μετόχους και από το Διοικητικό μας Συμβούλιο και αυτό επετεύχθη από ε, τις υπηρεσίες μας αλλά κυρίως από την Αντιπροεδρία της Τράπεζας. Ε, ο κ. Βεντούρ που εδώ είναι αυτός που ακούραστα δούλεψε για την νέα ενεργειακή πολιτική της Τράπεζας που, χρησιμο... συμπεριλάμβανε βέβαια την, την πάυση χρήσης των ορυκτών καυσίμων. Φαντάζεσαι τι αντίσταση βρήκε και Έπειτα, η υπεύθυνη αντιπρόεδρος ε, για τις κλιματικές αλλαγές, που θα είναι και η συνομιλήτριά σας, είναι ήδη όμως στη Μαδρίτη, ε, λόγω της COP25. Έχουμε και τον ε, κύριο Χαϊόλ που βεβαίως ε, έχει τις φιλοδοξίες για να συνδυάσει τη χρηματοδότηση με τα κλιματικά θέματα και πιέζει για αυτό το θέμα στην τράπεζα. Σας ευχαριστώ, τους ευχαριστώ πάρα πολύ και βεβαίως Κύριε Πρόεδρε, εάν οι ερωτήσεις που υποβληθούν αργότερα ε, δεν είναι της άμεσης αρμοδιότητάς μου, θα δώσω απευθείας το λόγο στους ε, δύο αντιπρόεδρους που, είναι, με συνοδεύουν. Αυξήσαμε, τις φιλοδοξίες ε, την περασμένη εβδομάδα μέσω του δικού σας ψηφίσματος για τις κλιματικές αλλαγές και το εκτιμώ όλος ιδιαίτερος. οι 4.000 υπάλληλοι της ΕΤΕΠ το εκτιμούν ιδιαίτερα γιατί στις 14 Νοεμβρίου αποφασίσαμε το κλίμα να γίνει η δική μας πρωτοβουλία. Εμείς θα σπάψουμε να χρηματοδοτούμε ε, project όπου δεν περιλαμβάνεται η μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων και θα χρηματοδοτούμε project που έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Από την εμπειρία μου πριν από μερικά χρόνια που εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι στηρίξαμε την ανάπτυξη, το ίδιο θα κάνουμε και τώρα και πιστεύω πως οι υπόλοιπε τράπεζες θα ακολουθήσουν. Οι στόχοι είναι σαφείς. Πρώτον, θα αυξήσουμε το μερίδιο των κλιματικών δράσεων και της χρηματοδότησης αυτών για την κλιματική βιωσιμότητα, να φτάσουμε στο, 25, ε, ε, στο 50% η τράπεζά μας λένε ορισμένοι ε, ότι θα πρέπει να γίνει κλιματική τράπεζα. Μα είμαστε όμως εδώ και πάνω από 25 χρόνια. Είμαστε ισχυρότεροι κατά πολύ ε, στον τομέα του κλίματος και έχουμε καλωσορίσει ήδη τα projects. Έχουμε, είχαμε ήδη 50% της χρηματοδότησης για κλιματικά project και σκοπεύουμε να φτάσουμε και πολύ πάνω από αυτό το ποσοστό. Το 2020 έχουμε να χρηματοδοτήσουμε ένα τρεις ε, σε τέτοια project ε, και μέχρι το 2030. Όταν ανακοίνωσα αυτό το νούμερο στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, το ανακοίνωσα όχι πολύ βέβαιος, αλλά αυτό ήταν πριν εγκριθεί από τις αρμόδιες ε, τα ε, όργανα της τράπεζας όμως τελικά συμφωνήθηκε. Ευθυγραμμίζουμε τις δραστηριότητές μας και μέχρι το τέλος του 2020 με τους στόχους του Παρισιού. Αυτό είναι κομμάτι του προγράμματος, γιατί αν δεσμευτείς να κάνεις 50% ε, δανεισμό για το κλίμα, δεν πρέπει να επιτρέπεται με το υπόλοιπο σου 50% να καταστρέφεις το κλίμα. Άρα λοιπόν, ή τους στόχους που έχεις επιτύχει μέσω της ε, κλιματικής σου χρηματοδότηση. Δηλαδή 50% με ήσυχη τη συνείδηση και 50% με ανήσυχη συνείδηση ε, δεν είναι καλή λύση. Αυτό σημαίνει πως επιγόντως πρέπει να υπάρχει σαφήνεια και διαφάνεια στο κομμάτι της χρηματοδότησης. Σε τα πράσινα μπον, ε, ομόλογα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, αφού εφευρεθήκαν πριν από κάποια χρόνια. Τότε μας πέρασαν για τρελούς. Αλλά ήταν τότε πιστεύω πολύ θαραλέο από πλευρά των προκατόχων μας. Ε, ε, αυτό το οποίο όμως κατέστησε αφές και πολύ σύντομα ήταν ότι πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες για το τι είναι ένα πράσινο ομόλογο. Δεν μπορείς να πάρεις ένα χαρτί και να το ονομάσεις πράσινο ομόλογο. Οι επενδυτές πρέπει να καταλάβουν και να γνωρίζουν ε, τι γίνεται με τα χρήματα, τι κάνεις με τα χρήματα που σου εμπιστεύονται. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, λογοδοσία και βιωσιμότητα. Και αυτό πρέπει να ελέγχεται και να υπάρχουν και διεθνή κριτήρια για το τι είναι πράσινη επένδυση. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ με τους εμπειρογνώμονές μας, αλλά συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα πολύ σταθερό πλαίσιο για τους ορισμούς. Το, οι πράσινες απάτες να σταματήσουν, η, το ξ, πράσινο ξέπλυμα, greenwashing. Και αυτό είναι κίνδυνος, όχι μόνο απέναντι στους πολίτες, γιατί χάνουμε την αξιοπιστία μας και μπορούμε να μην πιστεύουν ποιες κλιματικές πολιτικές. ε, ε, ε έχει να κάνει και με την εμπιστοσύνη των επενδυτών. αν ε, ε, ε, δεν καταλάβουν ότι τι κάνουμε με τα χρήματά τους, πάλι χάνουμε την αξιοπιστία μας. Γι' αυτό πρέπει να σταλεί ισχυρό μήνυμα στη Μαδρίτη, όπως η Ένωση είναι ο, ο κύριος αγωνιστής παγκοσμίω για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Και αυτό επίσης σημαίνει ότι μέσω της ταχείας ανάπτυξης της απαραίτητη τεχνολογίας με άλματα τεχνολογικά θα είμαστε στην πρωτοπορία για το ολόκληρο τον κόσμο. Εάν ε, ε, ε, συνεχίσουμε να χάνουμε την ανταγωνιστικότητά μας διότι δεν κάνουμε αρκετά με καινοτομία, τότε θα είναι πολύ προβληματική η κατάσταση. Εδώ και 15 χρόνια υπάρχουν χαμηλότερες επενδύσεις από ό,τι στους ανταγωνιστές μας για την κοινοτομία. Και δεν πρόκειται για ε, ε, ε, κάτι το οποίο είναι πάρεργο, όχι, είναι η βασική μας πολιτική. Πρέπει να συμβάλλουμε στην Πράσινη Συμφωνία. Πιστεύω πως πρέπει να, οι επενδύσεις να είναι κλιματικά ουδέτερες, να επιτύχουμε τους στόχους του Παρισιού, αλλά δυστυχώς οι δημόσιοι πόροι είναι λιγοστοί. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα μπορεί να κινητοποιήσει ιδιωτικέ επενδύσεις γιατί μπορεί να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε ρόλο κλειδί για το μελλοντικό ε, ταμείο ε, ε, βιώσιμων επενδύσεων. Επίσης θέλουμε να παρέχουμε υπηρεσίες ε, για να στηρίξουμε την Κομισιόν ε, τις πολιτικές τις γνωρίζουμε πολύ καλά πως η μεταβασή που χρειάζεται για να επιτυχθούν οι στόχοι του Παρισιού θα επηρεάσει ε, κάποιους τομείς και κάποιες περιοχές περισσότερο από ό,τι άλλες και εμείς δεσμευόμαστε να χρηματοδοτήσουμε τη μετάβαση εκεί ε, έτσι ώστε κανείς να μην μείνει πίσω. Μία νέα ενεργειακή πολιτική ήδη προτείνει μέτρα για την ανάπτυξη ενός πακέτου για την ενεργειακή μετάβαση, όπου περιλαμβάνεται η δυνατότητα κατ' εξαίρεση να χρηματοδοτηθεί μέχρι το 75% αντί 50% των, των κόστος των επιλέξιμων project, εφόσον η χώρα για την οποία πρόκειται, ε, πλήττεται περισσότερο από την ενεργειακή μετάβαση. Το θέμα όμως της ενεργειακής μετάβασης δεν αφορά μόνο ανανεώσιμη ενέργεια και ενεργειακή απόδοση, αλλά και νέες οικονομικές προπτικές, ανάπτυξη και δουλειές. Γιατί βεβαίως μέσω της μετάβασης θα χαθούν θέσεις απασχόλησης και ο κόσμος αυτός θα χρειαστεί νέες θέσεις. Και ε, αν και πρέπει ε, κάποιος που δούλευε ας πούμε σε ορυχείο να μπορέσει να εργαστεί και στο ψηφιακό κόσμο αργότερα και αυτό δεν γίνεται μέσα σε ένα χρόνο. Οι φιλοδοξίες είναι λοιπόν μεγάλες, ο όμιλος ΤΕΠ, δηλαδή η ίδια η τράπεζα και οι, και, και οι ε, της εργαζόμαστε ώστε να αποδώσουμε μέχρι το 2025 όπου θα σας παρουσιάσουμε το project μας ε, προσεχώς. Η Κλιματική Τράπεζα ε, ΕΤΕΠ και ο δικός χάρτης μέχρι το 2025 ενισχύει την κλιματική στρατηγική η οποία είναι υπό αναθεώρηση γιατί εγκρίθηκε το 2015 ενώ έχει σημειωθεί πολύ σημαντική πρόοδος από, από τότε ε, και ε, έχουμε προσαρμοστεί στις δεσμεύσεις που αναλάβαμε στο Πορίσι πριν από τέσσερα χρόνια. Εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε στενά, συνεργαζόμαστε μάλλον στενά με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς της Βρυξέλλες και το Στρασβούργο γιατί είναι προφανές ότι οι δραστηριότητες της τράπεζάς μας πάντοτε αποτελούνται από ένα, τριγωνικό, ένα τρίγωνο συνεργασίας, δηλαδή δανεισμός, έλεγχος στις πόρους της Ένωσης και συμβουλευτικός ρόλος. Όλα αυτά ε, μαζί απαιτούν συνεργασία με εσά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και βέβαια τη στήριξη των ίδιων των κρατών μελών όταν πρόκειται για το μέλλον ε, του προπολογισμού τη Ένωση. Και γι' αυτό και πρέπει να γνωρίζουμε τι περιλαμβάνει ε, το Πράσινο Σύμφωνο πέρα από το πακέτο δίκαιη μετάβαση. Μέχρι στιγμή είναι απλώ ένα προγραμματικό τίτλο. Τι επόμενε εβδομάδε ελπίζουμε πω θα ανακαλύψουμε περί τίνο πρόκειται με τη στενή συνεργασία μα με τον Φράντζα Τίμερμαν θα πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το πράσινο σύμφωνο. Γιατί μπορεί να μιλάμε για ένα όραμα, Αλλά ορισμένοι μπορεί να γελάνε μαζί μας γιατί πιστεύουν ότι χρειάζεται, χρειαζόμαστε ψυχίατρο επειδή έχουμε, βλέπουμε οράματα. Αντιθέτω, εμεί πιστεύουμε ότι πρέπει να δώσουμε σάρκα και οστά στο Πράσινο Σύμφωνο και το δίκαιη μετάβαση και το Ταμείο μάλλον δίκαιη μετάβαση. και μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι θα έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτού. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα και βεβαίω, είμαστε στη διάθεσή σα να απαντήσουμε σε ερωτήσει. και αν δεν μπορέσουμε να τι απαντήσουμε όλε στον περιορισμένο χρόνο που έχουμε σήμερα θα σα ε, απαντήσουμε ατομικά, προσωπικά στον καθέναν από εσά ε, Σα διαβεβαιώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Το μικρόφωνο φαίνεται να δουλεύει τώρα, οπότε ξανααλλάζουμε θέσεις. Seems to be working. Okay. Φαίνεται ότι λειτουργούν τα μικρόφωνα τώρα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τους συντονιστές από το ΕΛΚ. Ο Πέτερ Λίζη το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε έχω Αναφερθήκατε σε κάποια νούμερα και είπε και η καγκελάριος ε, όποιος έχει οράματα πρέπει να πάει στο γιατρό. Αλλά χρειάζονται παρόλα αυτά τα οράματα και Ελπίζουμε να έχει το ισχυρό αυτό όραμα για την ουδετερότητα του κλίματος η κυρία Φόντερ Λάιεν. Το είπε άλλωστε και το έχει υποστηρίξει, αλλά δεν είναι αρκετό το όραμα. Πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένες δράσεις. Η δίκαιη μετάβαση για μας το ΕΛΚΑ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πράγματι θα πρέπει πλέον να βάλουμε ε, σάρκα στα οστά, μπορώ να το θέσω έτσι σε ό,τι αφορά ε, την απομάκρυνση από τη χρήση του άνθρακα. Έχω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις προς εσάς. Ε, την τελευταία εβδομάδα με πολύ μεγάλη πλειοψηφία δεχθήκαμε αυτή τη δέσμευση της ε, ΤΕΠ και την μεταστροφή της σε επενδύσεις φιλοπεριβαλλοντικές. Τα unabated fossil fuels λέτε, δεν θα τα στηρίξετε. Τι θα πει αυτό βλέπετε κάποιες δυνατότητες για την ε, δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα για περαιτέρω στήριξη αυτής της ε, τεχνολογίας. Δεύτερη ερώτηση, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο τι θα γίνει ε, με τη χρήση του αερίου ως μεταβατική τεχνολογία σε συνδυασμό με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Νομίζουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο σε κάποια κράτη-μέλη, δεν είναι ο στόχος για το 2050, όμως αν λάβουμε υπόψη, παράδειγμα την Πολωνία και την κατάσταση με τον άνθρακα, υπάρχει πάρα πολύ άνθρακα πολύ λίγο αέριο ε, με τις ανανεώσιμες και νομίζω ότι είναι καλή η επένδυση αυτή και ελπίζω να μπορέσετε να την ενισχύσετε και περαιτέρω. So for SND, uh, to Mohamed Shahin. Mohamed Shahid από τους Σοσιαλιστικούς Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Δόκτωρ Χόιερ, σας ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγική παρέμβαση. Εμείς χαιρετίζουμε ω σοσιαλιστές και δημοκράτες τη μετάβαση ε, της ΕΤΕΠ σε μια τράπεζα έστω εν μέρη πιο φιλοπεριβαλλοντική. Τι εννοείται με χαμηλές εκπομπές αερίων ε, μας ε, ανησυχεί κάπως και μας ενδιαφέρει να το διευκρινίσετε όπως είπε και ο κύριος Λίζ. Οι επενδύσεις για το ορυκτά καύσιμα. Είπατε ότι αν είναι αμύωτες δεν τη στηρίξετε. Τι γίνεται με την πράσινη ταξινόμηση. Είπα το 5% των επενδύσεων της ΤΕΠΑ θα είναι πράσινες επενδύσεις και το 50% θα ε, αφορούν άλλους κλάδους. Πού θα πάνε αυτές οι επενδύσεις. Μήπως αυτές θα αντιβαίνουν τελικά τους στόχους της Συμφωνίας των Παρίσιων για το κλίμα. πέραν αυτή τη συζήτηση, δηλαδή για την πράσινη ταξινόμηση, μήπω θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση για την καφέ ταξινόμηση. Και αν αυτό θα βοηθήσει βέβαια και τι επενδύσει σε ΤΕΠ. For Νίλ Στόρβαλ για του ε, εκ του Ευχαριστώ, Πασκάλ. Ε, λίγο σε κοράκι φέρνει φωνή μου σήμερα και όχι τόσο σε άνθρωπο και λυπούμε. Γι' αυτό ζητώ συγγνώμη, τέλο πάντων. Ε, μιλήσετε για την ουδετερότητα. Έχουμε διαφορετικά τεχνολογικά υλικά, οργανι, οργανώσεις, ε, κάποιες συμφορήσεις ε, κτλ. Για τις διαφορές για τα κτίρια, για, τα διάφορα, για τους διάφορες κλάσεις του τα πράγματα δεν είναι πάντα τα ίδια. Υπάρχουν διαφορές. Και υπάρχουν και διαφορετικοί επενδυτικοί κύκλοι. Και άλλες προϋποθέσεις και όροι υπάρχουν, βιοποικιλότητα κτλ. Η τράπεζα θα πρέπει να μπορέσει κατά κάποιο τρόπο όλα αυτά να τα συμφιλιώσει, όλες αυτές τις διαφορετικές πτυχές. Σαν ένα καλλιδοσκόπιο δηλαδή, φανταστείτε το. Σαν να το στρέφει ο χρόνος και όταν το στρίβει ε, δίνει τελείως διαφορετική εικόνα. Πολύ απλό ερώτημα. Πώς θα να αντιμετωπίσετε. Όλα αυτά τα πολύ σοβαρά και ενίοτε μεταξύ τους ε, αντικρουόμενα ζητήματα. Ευχαριστώ. Για τους πρασίνους, ποιος έχει το λόγο, εσείς. Um, ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ, κύριε Χόιερ. Και εμείς οι πράσινοι θεωρούμε, ο κύριος Μπλός, ότι η ΕΤΕΠ κάνει ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση, ένα μεγάλο άλμα μάλιστα θα το χαρακτήριζα, αλλά έχουμε και εμεί κάποιε απορίε για τον τρόπο που θα προτιθέσετε να εφαρμόσετε όλα αυτά τα όσα αναφέρετε. Μιλήσατε για έναν οδικό χάρτη καταρχά. Θα μπορούσατε ίσω να μα εξηγήσετε τι εννοείται ακριβώ και ποια είναι τα ε, συγκεκριμένα βήματα για να πετύχουμε το στόχο του 50%. Με τι χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση άλλων δανειοληπτικών πολιτικών στον τομέα των μεταφορών. Και η ευθυγράμμιση που είπατε με τους στόχους των Παρισίων, πώς την εννοείται ακριβώς, και πώς δεν θα προκληθεί ζημία. Δανειοδότηση του αερίου. Έχουμε μια λίστα ε, που συνεχίζει να χρηματοδοτείται και το ίδιο θα ισχύει μέχρι το 2024, αν κατάλαβα καλά. Τι γίνεται με τα συστήματα θέρμανσης και τα λοιπά. Έχουμε κάποιες ε, απομονωμένες ε, κάπως ε, επενδύσεις μέσα σε αυτό το χαρτοφυλάκιο. Τι θα κάνετε με αυτό. Και σε ό,τι αφορά τον ορισμό του low carbon gas, μήπως το ρηκτό αέρα θα συνεχίσει να το επενδύετε, να επενδύετε σε αυτό μάλλον δυνάμει ακριβώς αυτού του ορισμού. Και τι γίνεται με αυτήν την κλιματική στρατηγική, την οποία αναθεωρείται. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Τι άλλα μέτρα, τι στόχοι συγκεκριμένοι υπάρχουν για την αναθεώρηση αυτής της στρατηγικής της ΕΤΕΠ για το κλίμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για το ECR. Αλεξάνδρου Βόντρα. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση πολύ συγκεκριμένη, αλλά θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε και ως γενική προσπάθεια να την θέσω στην Ολομέλεια πριν δύο εβδομάδες όταν ήταν οι συναδελφοί σας ε, εδώ αλλά δεν έλαβα κανένα είδου απάντηση. Εγώ είμαι από την Πράγα, στη Τσεχική Δημοκρατία. Παραδοσιακό σταυροδρόμι ε, που συνδέει το Βερολίνο με τη Βιέννη, τη Φραγκφούρτη με τη Βαρσοβία. Δεν έχουμε τελειώσει το δακτύλιο της Πράγας, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση μέσα στην Πράγα, λόγω των φορτηγών, των αυτοκινήτων και έχουμε ένα Δήμο του οποίου ηγούνται οι πειρατέ ε, που είναι μέλη του Πράσινου Κόμματο εδώ και υποσχέθηκαν ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα χρηματοδοτήσει ολόκληρο το δακτύλιο τη Πράγα. Και ε, εδώ έχω να κάνω την ερώτησή μου. Αν αυτό ο δακτύλιο ολοκληρωθεί, θα βελτιώσει εντυπωσιακά την ποιότητα του αέρα στην ε, πρωτεύουσα τη χώρα μου αλλά δεν πρόκειται ταυτόχρονα να συμμετέχει κατά κανένα τρόπο στους, στην επίτευξη των στόχων του Παρισιού. Απλά δηλαδή τα αυτοκίνητα θα παρακάπτουν την πόλη. Θα βελτιωθεί δηλαδή η ποιότητα του τοπικού αέρα, αλλά δεν θα συμβάλλουμε στην ποιότητα γενικότερα του αέρα. Στο νέο Transform EIB, στη νέα τράπεζα επενδύσεων, την οποία θα, που θα αλλάξει μορφή, θα υπάρξει κάποιο κονδύλιο τέτοιο για τέτοιου είδου επενδύσει. Θα είναι επιλέξιμε αυτέ οι επενδύσει για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για το ID και ζητώ συγγνώμη για την αλλαγή, αλλά δεν ήσασταν ε, στη λίστα Σιλβία Σαρτώνε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Χόιερ. Κύριε Χόιερ, όπως διάβασα, προτίθεστε να επενδύσετε ένα τρισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2030. Αυτό το νούμερο ε, έχει προγραμματίσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κλιματική ιστερία που έχει καταλάβει ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για σας το Green Deal είναι το μόνο πραγματικό εργαλείο για να αποφύγουμε να πεθάνει όλος ο πληθυσμός της γης. Είναι κάτι σοβαρό, τέλος πάντων. Και η ερώτησή μου είναι, αν όπως λέει η Γκρέτα, είναι κατεπήγον ο κίνδυνος αυτός μαζικής καταστροφής. Πώς είναι δυνατόν να ε, βγάζουμε επενδύσεις ε, δημόσιες από την κλιματική αυτή, από το κλιματικό κίνδυνο. Δηλαδή, να εξηγήσω, αν πάτε και λέτε ότι θα πεθάνουμε όλοι, και αυτό από την προτεραιότητα, πώς ξαφνικά βάζετε ως δέσμευση ε, το να τηρούμε την ισορροπία στον προπολογισμό. Ούτε ιδεολογικά δεν προβλέπετε καμία εξαίρεση. Μου φαίνεται ότι μας κάνετε πλάκα. Το να τη μετατρέψετε την τράπεζά σας σε κλιματική τράπεζα είναι μια απόπειρα, μια απόπειρα απελπισμένη να σώσετε το δικό σας χρηματοοικονομικό σύστημα, το χρηματοπιστωτικό σας σύστημα. Φαίνεται εσείς να θέλετε περισσότερο να εξυπηρετήσετε τους μεγάλους επενδυτές των τραπεζών και τις μεγάλες επενδύσεις παρά να προστατέψετε του πολίτε και να καλύψετε τις πραγματικές του ανάγκες. Μπορείτε λοιπόν να μου εξηγήσετε πώς ε, συνδυάζεται η, αφενός η βούληση ε, καταπολέμησης ε, του κινδύνου αυτού που μπορεί όλοι να πεθάνουν λόγω του κλίματος που επιδεινώνεται καθημερινά αφετέρου να προβλέπετε συγκεκριμένα ε, ποσοστά με πολύ μεγάλη ακρίβεια και περιορισμού για το πόσο τα κράτη μπορούν να επενδύσουν σε αυτόν τον πολύ σημαντικό κλάδο. Thank you. The last uh, coordinator... Ευχαριστώ. Τελευταίο ε, συντονιστή, ε, Μόντι και την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Χόιερ για την παρουσίαση αυτή. Σε γενικές γραμμές είναι πολύ καλή απόφαση αυτή. για την υποστήριξη επενδύσεων ε, απαλλαγή ε, από τον άνθρακα. Και έτσι έχουμε επιτέλους μια χρηματοδότηση ε, που υποστηρίζει τους κλιματικούς στόχους. Το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ στενό. Έχουμε τις δημόσιες συμβάσεις και τις δημόσιες επενδύσεις στα κράτη-μέλη που αντίκυνται στους κλιματικούς στόχους και αυτό που θέλει σπατάλη χρημάτων. Έχω δύο ερωτήσει. Μία για το φυσικό αέριο που έθεσε και ένα συνάδελφο και η δεύτερη για την ενεργειακή απόδοση. Εσείς ε, αναφερθήκατε στους στόχους του 2050, που είναι ο συνολικός στόχος, ο γενικός στόχος. Εμείς θεωρούμε ότι ο στόχος του 2030 είναι ο σημαντικότερος. Θα χρειαστεί λοιπόν ένας οδικός χάρτης για να τον επιτύχουμε. Διαφορετικά θα μας ξεφύγει. Ε, λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρος Αλλά οι στόχοι δεν ε, βασίζονται ακόμα σε επιστημονικά στοιχεία, ούτε είμαστε ακόμα στο, έχουμε φτάσει στο σωστό επίπεδο. Αυτά που ακούμε για το Green Deal και για το δέσμη μέτρο για την πράσινη οικονομία, όλα αυτά ακόμα δεν ε, χαρακτηρίζονται από αρκετά φιλόδοξους στόχους. Δεδομένου αυτού δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι είμαστε πρωτοπόροι ούτε ηγέτες στον κλάδο. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω για τα, φυσικά, για τα, συγγνώμη, για τα καυσαέρια, όχι για τα φυσικά αέρια, για τα καυσαέρια. Θεωρείτε ότι το CCS είναι πραγματικά η λύση? Θεωρώ ότι οι λύσει ευρεία κλίμακα δεν υπάρχουν διαθέσιμε. Οπότε, τι γίνεται με τα καύσιμα ε, και τι χαμηλέ εκπομπέ ε, καυσαερίων δεν θα ήταν καλύτερα να περάσουμε κατευθείαν σε καθαρές, πραγματικά καθαρές ε, πηγές ενέργειας. Το φυσικό αέριο μπορεί να είναι μια μεταβατική λύση. Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά την ενεργειακή απόδοση, κάτι που πρέπει να υποστηρίξουμε, αλλά ποια είναι τα κριτήρια που θα μας βοηθήσουν να διασφαλίσουμε ότι οι επενδύσεις σε θέματα ενεργειακής απόδοσης θα λαμβάνουν υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής κτηρίων και των υλικών. Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε, πάμε και στις άλλες ερωτήσεις, γιατί αλλιώ δεν θα προλάβετε να απαντήσετε. Κλείνω λοιπόν τον κατάλογο εδώ. Έχω περίπου 9 επιπλέον ομιλητές. Παρακαλώ, περιοριστείτε στο ένα λεπτό για τις ερωτήσεις σας, αλλιώς δεν θα λάβετε απαντήσεις. Ζητώ συγγνώμη. Έχετε μεγάλη επιτυχία αλλά μετά ε, πρέπει να μην καθυστερήσουμε με την ψηφοφορία. Ε, ΕΛΚ λοιπόν, η κυρία Μαρία Σπυράκη. Thank you, Chair, for giving... Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Χόγερ που ήρθατε εδώ για αυτή τη συζήτηση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Δύο ερωτήσει πολύ σύντομα. Πρώτον, στην χώρα μου, στην Ελλάδα, έχουμε δύο περιοχέ σε μετάβαση. Η Δυτική Μακεδονία είναι η πρώτη και η δεύτερη είναι η πόλη της Μεγαλόπολης. Ήθελα να σας ρωτήσω, ειλικρινά πείτε μου, έχετε να μας προτείνετε τίποτα στις τοπικές αρχές για να αρχίσουν ε, να παρέχουν ε, νέα επιλέξιμα έργα για ε, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και δεύτερον η ερώτηση που αφορά τη χρήση φυσικού αερίου ως μεταβατικής πηγής. Ήθελα να σας ε, ρωτήσω στο ίδιο πλαίσιο, εάν αυτές οι σε μετάβαση περιοχές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το φυσικό αέριο με διευκόλυνση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αυτό θα ήταν δυνατόν μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Σπορέκ, μαζί με την έγκριση της νέας ενεργειακής πολιτικής το 14 Νοεμβρίου, οι διευθυντέ της Τράπεζας Επενδύσεων ενέκριναν μια νέα στρατηγική που αυξάνει τη χρηματοδότηση για την κλιματική δράση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ώστε να φτάσει στο 50% των δραστηριοτήτων το 2025 και στη συνέχεια. Μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είχε στόχο 25% που είχε αφοσιωθεί στο έργα κλιματικής δράσης μόνο. Και αυτή η τελευταία αύξηση έως το 50% δεν είναι μόνο ποσοστία, αλλά και σε κλίμακα. Δεν περιλαμβάνει μόνο δηλαδή την κλιματική διάσταση των έργων, δηλαδή μόνο την οριζόντια διάσταση, αλλά και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Κάτι ξεχωριστό ε, ως κλάδος έργων, κατακόρυφο. Με την υπάρξη μεθοδολογία τη τράπεζα δεν είναι δυνατό σήμερα να υπολογίσουμε πώ θα επιτευχθεί ο στόχο αυτό. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι ποιο είναι ο νέο ακριβή στόχο για την κλιματική δράση και ποια μεθοδολογία θα ακολουθηθεί για τον υπολογισμό του. Thank you for renew. Ευχαριστούμε για το Renew, ο κύριος Γιάνν Χουίτεμα. Δεν είναι εδώ, Μάρτιν Όισιτς. Ε- Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Πολύ ενδιαφέρουσα. Ήθελα να ρωτήσω αυτή η πολιτική δανειοδότηση, ε, που είναι καλό βήμα μπροστά θεωρώ πώς μπορεί να συμβάλλει στη σταδιακή εξέλιξη στην Ευρώπη. Εγώ έρχομαι από μια περιοχή που συχνά εξαρτάται πολύ ε, από τα καύσιμα, από τα ορεκτά καύσιμα εξαρτάται επίσης ε, και πάρα πολύ από βιομηχανίες ε, έντονα ενεργοβόρους. και ήθελα να μάθω αυτή η δανειοδοτική πολιτική θα βοηθήσει να υπερβούμε ε, να μετα... υπερπηδήσουμε το τεχνολογικό χάσμα και να μπορέσουμε να σημειώσουμε κάποια εξέλιξη. Ευχαριστώ για τους πρασίνους. Η κυρία Παύλου ευχαριστώ πολύ. Ε, πρόεδρε, και ευχαριστούμε κύριε Χόγερ που είστε εδώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ. Η βιοπικιλότητα ως κρίση Παραβλέπετε συχνά σε σχέση με τη γενικότερη κλιματική κρίση. Θα με ενδιαφέρει να μάθω ε, τι είδους έργα θα θέλει να χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε αυτό το τομέα πολιτικής. Ε, θεωρείτε ότι θα χρηματοδοτήσετε έργα διατήρησης ή γεωργικά, για παράδειγμα έργα που ενισχύουν τη βιοπικιλότητα ή έργα όπω οι πιο πράσινε πόλει ή ε, η βιοπικιλότητα στι πόλει. Θα μπορούσατε να με διαφωτίσετε λίγο, παρακαλώ. Thank you for ECR. Ευχαριστούμε για το ECR, η κυρία Ζαγιουσκά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ και έχω μερικές ερωτήσεις. Βρίσκομαι... Ε, η τράπεζα που διευθύνεται είναι ένας ανεξάρτητος ε, οργανισμός, έχει νομική υπόσταση, νομική προσωπικότητα και διαχειρίζεται δημόσια και ιδιωτικά χρήματα. Και η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξής. Η συνεργασία με την ε, Επιτροπή η οποία θεω, ελπίζουμε ότι σύντομα θα μας παρουσιάσει κάποια οδηγία και κάποιες αρχές. Μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο δυνατά στο μικρόφωνο σας για τους μεταφραστές, παρακαλώ. Thank you E, to e, e, pierwsze, pytanie, jak την ερώτησή μου, πώς θα γίνει η συνεργασία με την Κομισιόν. Πώς φαντάζεστε ότι θα διαχειριστείτε αυτά τα ε, κολοσσιαία ποσά. Ε, ε, θα περίμενα λοιπόν να μας πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο, πιο ακριβές. Δηλαδή, ε, ακόμα περιμένω να μας πείτε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και η δεύτερη μου ερώτηση αφορά το φυσικό αέριο. Πράγματι, εμείς ανησυχούμε ε, από κάποιες φήμες που κυκλοφορούν ότι η τράπεζα ετοιμάζεται να απορρίψει τη χρηματοδότηση έργου που θα σχετίζονται με το φυσικό αέριο. Αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερω, διότι η Πολωνία επενδύει πολύ σε έργα φυσικού αερίου. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε για την ΚΟΕ. Thanks, Chair. Um, Dr. your, um... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριο Βουάλλα, η τελική σα πολιτική διατηρεί την ρήτρα αναθεώρηση. Δεν έχω το αρχικό σχέδιο που θα επιτρέπει να αντιληθούν χρήματα, να μπουν χρήματα στα έργα φυσικού αερίου στην Ιρλανδία, το οποίο θα μας κάνει να εισάγουμε ε, ε, φυσικό αέριο σχιστολιθικό αέριο από την Αμερική για δεκαετίες. Ο αντιπρόεδρος που κάθεται εκεί, ο Άντριου, ε, στα αριστερά σας είπε πρόσφατα σε μια συνέντευξη ότι η AB θα συνεχίσει ε, να χρηματοδοτεί ε, τα έργα φυσικού αερίου μετά το 2021 εφόσον τηρούν τα αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα. Μπορείτε να μας αναλύσετε. Επίσης λέει ότι γενικά θα εγκρίνεται ηλεκτροπαραγωγικά έργα που θα εκλείουν λιγότερο από 250 ε, κυβικά μέτρα ανά ώρα. Όλα αυτά είναι πληροφορίες από μια ομάδα τεχνικών επιρρογνωμόνων. Ε, σύμφωνα με την ομάδα τεχνικών επιρογνωμόνων, δεν θεωρούνται ε, ε σωστές δραστηριότητες αυτούς του παραγωγής φυσικού αερίου διότι εκλείουν πολύ περισσότερο. Οπότε δεν θεωρούνται ότι συμβάλλουν επαρκώς ε, στην μετριασμό των κλιματικών αλλαγών. Οπότε δυόμιση φορές παραπάνω είναι το όριο που έχετε θέσει εσείς σε σχέση με αυτό που επιτρέπετε. Μπορείτε να εξηγήσετε. Ευχαριστώ για τους τρεις τελευταίους ομιλητές για το ΕΛΚ και η κυρία Μπέντελε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Χοϊερ για την ε, παρουσίαση. Σε ποιο βαθμό θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν ήδη επιστώσεις ε, ε, για χρηματοδότηση κλιματικών στόχων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχει περίπτωση να ενταθούν αυτά τα μέτρα. Εγώ ερωτώ, ε, εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε αποφασίσει τα μέτρα σε θέματα αναπτυξιακής βοήθειας ε, να διπλασιάζονται όταν ε, υπάρχουν και μέτρα ε, κλιματικά στην επόμενη θητεία και φυσικά θέλουμε να υπάρχει προστασία του κλίματος διεθνώς και θέλουμε και περισσότερη συμμετοχή επίσης του ιδιωτικού τομέα. Ευχαριστώ. Thank you for le... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χόγερ, λέει ο κύριο ε, Είναι πολύ σημαντικές οι λύσεις ε, αυτές που βρίσκεται ε, η πορεία σας είναι να χρηματοδοτείτε πολύ σίγουρα προγράμματα για να μην χάσετε την αξιοπιστία σας. Όμως εκπλήσει κάπως αυτή σας η στάση γιατί είμαστε μπροστά σε μια αναπτυξιακή τράπεζα. Άρα λοιπόν πώς προτίθεστε να συνδυάσετε το τριπλό σας α, αυτή την μανία σας να διατηρήσετε το τριπλό α και τη χρηματοδότηση πράσινων project που είναι τόσο σημαντικά για το κλίμα αλλά που μπορεί να μην είναι τόσο σίγουρα επενδυτικά projects όσο άλλες επενδύσεις. Ευχαριστώ. Τέλος από το Renew. Έχω μία πολύ σύντομη ε, ε, ερώτηση. Ε, μάλλον να ξαναρχίσω, λέει ο κύριος Χουίτεμα. Οι πράσινε εταιρείε είναι, πιστεύω, η κινητήριο δύναμη για την καινοτομία. Πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα που θα δαπανίσει η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα θα πάνε στου σωστού ανθρώπου και στι μικρομεσαίε επιχειρήσει επίση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ε, ζητήσω να απαντήσετε όλες αυτές τις ερωτήσεις σε μάξιμουμ 15 λεπτά μίνιμουμ 10, μάξιμουμ 15 λεπτά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ γενναιόδορη η προσφορά σας. Σας ευχαριστώ. Ε, καταλαβαίνω τους ε, χρονικούς περιορισμούς. Κάτι αντιλαμβάνομαι. Είναι πολλές ερωτήσεις. Θέλω να προσπαθήσω να απαντήσω στο μέγιστο βαθμό. Αλλά παρακαλώ θυμίστε μου αν δεν λάβετε την απάντηση. Ε, και αλλιώ επικοινωνήστε με το γραφείο μου στις Βρυξέλλες. Αλλά γενικά. Ε, η κλίμακα αυτή των ερωτήσεων, το εύρο των ερωτήσεων και η τελευταία που ακούσαμε για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει δείχνει το εύρο δραστηριοτήτων που αναμένεται να επιτελέσει η τράπεζα. Είμαστε μια κλιματική τράπεζα, όπω είπαμε, και θα συνεχίσουμε να είμαστε αυτό. Θα είμαστε η κλιματική τράπεζα για πολύ καιρό. Και το κλίμα θα βρίσκεται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο. Ταυτόχρονα όμω αναμένουμε να δημιουργήσουν και θέσει εργασία οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ταυτόχρονα ε, προσδοκούμε να καταπολεμήσουμε και την απώλεια παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τους εμπορικούς μας εταίρους, επενδύοντας πολύ περισσότερο στην καινοτομία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μας αδυναμία. Ταυτόχρονα αναμένεται εμείς να συμβάλλουμε στο όραμα και στη φιλοδοξία του να είμαστε πρωτοπόροι παγκοσμίω και στο πλαίσιο αυτό να έχουμε μια στρατηγική αυτονομία. Για μένα ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που έχουμε ως φιλοδοξία τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να συμβάλλουμε λοιπόν σε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε διάφορες ομάδες στόχων, κλίμα, καινοτομία, ανάπτυξη και απασχόληση και κάποιους άλλους. Και πρέπει να διασφαλίσουμε να... ότι δεν θα πνιγούμε μέσα σε όλο αυτό το σύνολο φιλοδοξιών και στόχων, θα μπορέσουμε να συμφιλιώσουμε στόχους που αρχικά φαίνεται να είναι αντιφατικοί. Ας δούμε ένα ενδιαφέρον παραδείγμα στη γειτονία μας, στα Δυτικά Βαλκάνια. Ε, μια περιοχή που θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη προσοχή από πλευρά μας. Στα Δυτικά Βαλκάνια βλέπουμε ότι αυτέ οι χώρε. στο πλαίσιο της πορείας τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μια μορφή ε, πολιτικής συνοχής χρησιμοποιούν πάρα πολύ την καινοτομία. Αυτέ οι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων είναι πολύ φιλόδοξε σε θέματα καινοτομία και τα καταφέρνουν πολύ, στη, τουλάχιστον οικονομικά, σε αυτή την πορεία του προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί λοιπόν, ε, αυτό είναι ένα παράδειγμα συμφιλίωση των φιλοδοξιών μα. Και όπω είπα και στη Γενική Συνέλευση ε, των Εθνών και στο Παρίσι πρόσφατα και ε, την επόμενη εβδομάδα στη Μαδρίτη, θα πρέπει ό,τι κάνουμε να χαρακτηρίζεται από το κλίμα. Ο σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι δεν υπονομεύουμε τις κλιματικές μας επιτυχίες με τις άλλε μας δραστηριότητες. Δεν είναι εύκολο, διότι ορισμένε φορές εξάγουμε τα λάθο συμπεράσματα. Εγώ πιστεύω ότι σε ένα κόσμο στον οποίο θέλουμε να είμαστε οικονομική δύναμη και τεχνολογική, τεχνολογικά πρωτοπόροι, φανταστείτε, χρειαζόμαστε δίκτυα, δρόμους, σιδηροδρόμους, αεροπορικές γραμμές, λιμάνια. Δεν θα αλλάξει αυτό αλλά αυτό πρέπει να γίνεται βιώσιμα. Γι' αυτό δεν είμαστε ονειροπόλοι. Πιστεύουμε ότι οι επιτυχίες σε θέματα κλίματος και διατήρησης της φύσης πρέπει να εκτελούνται με τι υψηλότερες τεχνολογικές φιλοδοξίες και φιλοδοξίες σε θέματα καινοτομίας. Οπότε εκεί ήταν πολύ ενδιαφέρον ε, το ερώτημα για τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει αλματώδης ανάπτυξη. Το είπε ο συνάδελφος από την Πολωνία. Αυτό ισχύει και για την κατάσταση ενδοκινοτικά. Έχουμε περιοχές όπου χρειάζεται αλματώδης ανάπτυξη. Στην Αφρική είναι προφανές. Τα κίνητρα σε χώρες όπως το Καμερούν ή η Αιθιοπία είναι τεράστια. Βλέπετε ότι το κινητό τηλέφωνο αποτέλεσε επανάσταση για τις κοινωνίες τους. Προσέφερε πρόσβαση σε πληροφορίες, σε πληροφορίες για την υγεία, σε ασφάλειες, σε τραπεζικές δραστηριότητες, σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε τράπεζα ήταν πραγματικά αδύνατη. αποτέλεσε, κέντρισε την οικονομική δραστηριότητα, ε, τη δραστηριότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μικροεπιχειρήσεων, για ανθρώπου που δεν είχαν καμία πρόσβαση στι αγορέ καθόλου. Αυτέ οι εξελίξει λοιπόν έκαναν τεράστια διαφορά. Και η Αφρική χαρακτηρίζεται από αυτό, αφού παραμελήθηκε για πάρα πολύ χρόνο, τώρα σκέφτονται αντί να επενδύσουν σε χάλκινα καλώδια για τις τηλεπικοινωνίες, επενδύουν στις ε, ε, ε, επικοινωνίες, στις κινητές επικοινωνίες. Αυτό έγινε με τη δική μας υποστήριξη, αλλά μπορούμε να κάνουμε όσο μπορούμε να κάνουμε, όσο μας επιτρέπετε εσείς, τα μέλη του Κοινοβουλίου, αλλά και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής διστάζουμε να πάμε σε πάνω από 10% δανειοδότηση εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σε αναπτυσσόμενε χώρε. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Μετά από τη μεταναστευτική κρίση, και δυστυχώ η μεταναστευτική κρίση ήταν αυτό που ξύπνησε του Ευρωπαίου σε θέματα ε, αναπτυξιακών δυσκολιών. Τώρα καταλαβαίνουν τι σημαίνει η Αφρική ε, να έχει 4 εκατομμύρια ανθρώπου μέχρι τα τέλη. Ε, 4 δισεκατομμύρια ανθρώπου μέχρι τα τέλη του αιώνα και τι στρατηγικέ πρέπει Να ακολουθηθούν και ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την αναπτυξιακή βοήθεια. Η ανάπτυξη λοιπόν είναι άλλο ένα τομέα όπου θα πρέπει οι στόχοι μα να συνδυάζονται επιτυχώ. Αλλά είναι αυτονόητο. Οποιοδήποτε αναπτυξιακό έργο υποστηρίζουμε στην Αφρική, στην, Ανατολή, στην Νότια Αμερική, ε, στην Ανατολική μα γειτονία, πρέπει να πληρεί τα πρότυπα που εφαρμόζουμε και εμεί ε, περιβαλλοντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να είναι αποδεκτό. Και αυτό θα κατευθύνει τι δραστηριότητε μα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, στο δεύτερο μέρο των απαντήσεων μου, θα ήθελα να αναφερθώ στα χρησιμοποιητά ε, περιουσιακά στοιχεία που αναφέρθηκα, τα stranded assets. Αυτό είναι κλειδί. Ε, πολλοί άνθρωποι καλόβουλα και με πολύ ωραίες ιδεολογικές ε, ιδεολογίες για, το κλίμα τα λένε όλα αυτά, αλλά εγώ δεν είμαι τόσο ιδεολογός. Θέλω με τεχνολογία και ρεαλιστικά να επιτύχουμε τους κλιματικούς στόχους. Θέλω να επενδύσουμε σε περιουσιακά στοιχεία που δεν θα αποσβεστούν γρήγορα. Είναι σημαντικό αυτό. Όταν μιλάμε για μια επένδυση που έχει διάρκεια ζωή 40 χρόνια και εξίσου ότι σε 30 χρόνια έχει πεθάνει, αυτό είναι ανεύθυνη ε, ανεύθυνο banking. Φανταστείτε να συζητήσει κάτι τέτοιο με του επικεφαλεί των μεγαλύτερων εμπορικών τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών στην Ευρώπη που θα σε χρηματοδοτήσουν και αυτοί θα σα πούν το ίδιο. Θα σα πούν είστε τρελοί να μπείτε σε τέτοιου είδου επενδύσει αφού ξέρετε ότι θα αποσβεστούν. Οπότε από αυτή την άποψη το ζήτημα των αχρησιμοποιητών περιουσιακών στοιχείων των stranded assets μας αναγκάζει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Διαφορετικά η ανάγκη αυτή διαγραφής ε, που θα οδηγήσει σε ζημίες για την τράπεζα θα καταλήξει στην τσέπη του φορολογωμένου πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωση, Δεν αποτελεί λοιπόν επιλογή. Το τρίτο ζήτημα που θα ήθελα να συζητήσω είναι αυτός ο κύκλος ζωή. και ο σχετικό τρόπος σκέψης. Πράγματι έχουμε ένα χάσμα εδώ, αλλά αυτό ισχύει γενικότερα. Εμείς στην Ευρώπη δεν επενδύσαμε, δεν αρκετά από την αρχή όταν κάνουμε κάποιο επενδυτικό έργο για την προβλέψιμη συντήρηση του έργου αυτού, ώστε να φτάσει στο τέλο ε, το έργο αυτό του κύκλου ζωή του. Και αυτό οδηγεί σε ένα χάσμα και σε μείωση τη ποιότητα ε, ε, των υποδομών και πολλέ φορέ σε κάποιε καταστροφέ. Σε κάποιο βαθμό η γέφυρα που κατέρευσε στην Ιταλία θα μπορούσε να έχει γκρεμιστεί, να έχει καταρρεύσει οποιοδήποτε άλλο μέρο τη Ευρώπη. Μην απλανάστε. Είναι πολύ σημαντικό το να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα και σε θέματα επισκευή, αποκατάσταση και συντήρηση. Και σε ενεργειακά έργα, σε ορισμένε περιπτώσει, θα χρειαστεί κάποια στιγμή να αποσύρουμε κάποια ε, σε εγκαταστάσει που κοστίζουν υπερβολικά. Και το τελευταίο μου σχόλιο, και μετά θα δώσω το λόγο στου συναδέλφου μου για τι μεταφορέ και για τα θέματα τη ενέργεια. Θα ήθελα να σα πω ε, κάτι για τα ανθρακοριχεία. Έχουμε μεγάλε φιλοδοξίε. Είχαμε μια προπαρασκευαστική διάσκεψη εξαιρετική για την Χιλή, ε, συγγνώμη τώρα για τη Μαδρίτη φυσικά, με το συνασπισμό των Υπουργών Κλίματος ε, και στο Βατικανό με τον Πάπα. Μια εκδήλωση πάρα πολύ φιλόδοξη. Και εκεί κατέστησε πόσο σημαντικό θα είναι το θέμα για όλους μας. Και αυτό σημαίνει για μας ότι πρέπει να επικεντρωθούμε ακόμα περισσότερο σε αυτά που ήδη κάνουμε σε χώρες εκτός Ευρώπης. Αλλά η αναδάσωση η γεωργία είναι όλο και πιο σημαντική. Η φιλοδοξία μας για τους ωκεανούς εκφράστηκε μέσω της πρωτοβουλίας για τους καθαρούς ωκεανούς που αναλάβαμε πριν δύο χρόνια μαζί με μια εταιρεία από την Γαλλία και μια από τη Γερμανία και τώρα έχουμε και άλλους. Όλα αυτά θα τα εξελίξουμε περισσότερο. Και θα πάμε στο Κουνμίνγκ με μια φιλόδοξη ατζέντα. Και ανα πάσα στιγμή θα ερχόμαστε να σας αναφέρουμε εδώ πριν πάμε εδώ. Και λοιπόν να δώσω το λόγο στον Άντρου για τις άλλες ερωτήσεις, ξεκινώντας από την ενέργεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλές ήταν οι ερωτήσεις για τον ρόλο του φυσικού αερίου στη νέα ε, πολιτική μας, για την ενέργεια, για την ενεργειακή απόδοση, τον ρόλο του αερίου. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η δανειοδοτική πολιτική μα δεν απορρίπτει εντελώ το ρόλο του φυσικού αερίου στη μετάβαση στην ενεργειακή, αλλά λέμε ότι σύμφωνα με τους στόχους της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια, ο τομέας ε, του φυσικού αερίου θα πρέπει να ε, πάψει να χρησιμοποιεί άνθρακα, να γίνει unabated, και υπάρχουν νέες τεχνολογίες, υπάρχουν αυτά τα ε, ε, κονδύλια τα οποία παραμένουν απομονωμένα και αχρησιμοποιητά και πρέπει να προωθηθούν τεχνολογίες ε, που θα μπορούν να βοηθήσουν στην αλλαγή της τεχνολογίας ε, γιατί διαλείπουσα αιωλική και ηλιακή ενέργεια βοηθάει το να έχουμε συμπλήρωμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα, φυσικό αέριο. Τι θα πει αυτό βέβαια αυτό που προτείνουμε στο έγγραφό μας είναι ότι για την παραγωγή ισχύω οι νέοι σταθμοί θα χρησιμοποιούν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες, αλλά θα πρέπει να είναι 250 μιλιγκράμμ διοξιδίου του άνθρακα ανά κιλοβατόρα οι εγνές οριακές τιμές για την εκπομπή αερίων από το φυσικό αέριο. Και αυτά τα project μπορούν τρία πράγματα να κάνουν. χρησιμοποιήσουν τις διαθέσιμες τεχνολογίες τεχνολογίες, συνδυάζοντας θέρμανση και ισχύ και το πλεόνασμα χρησιμοποιείται για θέρμανση νερού, ιδίω ε, για τα αστικά συστήματα θέρμανσης. Είναι πολύ αποτελεσματική αυτή η τεχνολογία και μειώνει τις εκπομπές που σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας, με το διοξείδιο του δεύτερον με μείγμα ε, βιοαερίου, συνθετικού αερίου και στο μέλλον ε, πράσινου υδρογόνου σε αυτό το μείγμα ε, που χρησιμοποιούμε για την ε, παραγωγή ενέργειας. Και έτσι ε, θα έχουμε εκπομπές κάτω από το όριο των 250. Και το τρίτο είναι να υπάρχει συνδυασμός με την τεχνολογία συνδέσμευσης και αποθηκεύσης άνθρακα, που είναι μια πολύ δαπανηρή τεχνολογία και είναι σε πρόωρο, πρώιμο στάδιο ακόμη. Εμείς θέλουμε να δώσουμε και βοήθεια στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού, το έχουμε το Ταμείο Εξυγχρονισμού, το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκόσμια κτλ. Και θέλουμε όλα αυτά να τα καταστήσουμε πιο ενδιαφέροντα για τους επενδυτές. Γιατί έχουμε αυτό το πρότυπο 250 και όχι 100. The sustainable Το θέμα είναι να ορίσουμε τα πράσινα οικονομικά με αυτή την ταξινόμηση, την ταξινόμηση ότι δηλαδή έχει πολύ θετική συμβολή στην κλιματική δράση και τους άλλους περιβαλλοντικούς στόχους. Το πρότυπο το 250 είναι για την ευθυγράμμιση με τη Συμφωνία των Παρισίων που είναι πιο χαμηλό αυτό το πρότυπο που λέει δεν πρέπει να προκαλέσουμε βλάβη, όχι να έχουμε μια τρομερά θετική συνεισφορά για να πάρει την ταμπέλα της πράσινης ε, χρηματοδότησης, του πράσινου οικονομίας, αλλά να μην προκαλέσει μια Εκεί έχουμε αυτό το πρότυπο 250. Ε, οι ανανεώσιμες έχουν το 100 ως πρότυπο αν χρησιμοποιήσουμε συνδυασμένου σταθμούς ε, με 250, έχουμε ευθυγραμμιστεί με τη Συμφωνία των Παρισίων, αλλά δεν παίρνει την ε, ετικέτα του Green Finance. Και σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση, πολύ ενδιαφέρον ο τομέας αυτός, ένας τομέας που έχει παραγνωριστεί, ε, γιατί Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι προσφέρει πολύ μεγάλες δυνατότητες ε, για τη χρηματοδότηση από πλευράς ΕΤΕΠ και σύμφωνα και με τους στόχους τους κλιματικούς της Ένωσης, τα νούμερα τα ξέρουμε, 200 δις επενδύσεων ε, το χρόνο χρειάζονται για να επιτευχθούν οι στόχοι. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι μέχρι τα τέλη του 2020 όλα τα νέα κτίρια που χρηματοδοτούμε θα πρέπει να πληρούν την απέτηση για σχεδόν μηδενική ε, ενέργεια και μετά θα είναι υποχρεωτικό και θα χρειαστεί ένα νέο πρότυπο. Μια νέα διαδικασία λοιπόν για την Τράπεζα και την Κομισιόν για αυτό το νέο πρότυπο που δεν θα εστιάζει μάλλον μόνο στην ε, απόδοση του κτηρίου αλλά και στον κύκλο ζωής ε, στην ε, σωματωμένη απόδοση του κτηρίου σε ό,τι αφορά τον άνθρακα. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας. Έχουμε ξεπεράσει τα 50 λεπτά. Αυτό που είπατε ε, ότι θα μπορούσατε να ξαναέρθετε, το κατέγραψα και ίσως λάβετε πρόσκληση να ξανάρθετε για να μας πείτε για τη στρατηγική. Βέβαια θα ψηφίσουμε και σε δύο λεπτά εμείς ε, θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε και εσάς και την ομάδα σας. Τα ξαναπούμε σύντομα. So I'm going to switch to French for the voting session. Για την ψηφοφορία θα αλλάξω γλώσσα και θα τα λέω γαλλικά. Δεν το κάνω πάντα. Ή τέλος πάντων δεν θα μιλήσω γαλλικά όλη την ώρα. Ξεκινώ στα αγγλικά. Πρώτη ψηφοφορία. Έχετε την κάρτα ψηφοφορίας. Το πρώτο θέμα λοιπόν. The vote is open. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέραση ψηφοφορίας. Rejected. We move to second vote on imports of pet food from... Για το δεύτερο, τη δεύτερη ένσταση για τα, τις ζωοτροφές από την Σαουδική Αραβία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεν το βλέπετε από ό,τι φαίνεται. 58 ψήφοι κατά, 12 υπέρ. Να φαίνεται παρακαλώ και στην οθόνη από εδώ και πέρα, αν μπορείτε, το αποτέλεσμα. Όπως είπαμε, 12 υπέρ, 58 κατά. Και 71 είναι ψεφίσαντες. είχαμε και μία αποχή. Επόμενο θέμα, τρίτο. να άρχεται η ψηφοφορία. Συγγνώμη, συγγνώμη. Συγγνώμη, υπάρχει μια προηγούμενη ψηφοφορία για τη Φουκουσίμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Ah. So, uh, minus... 40 ψήφοι κατά, 30 υπέρ. Αποχή μία. Απορρίπτεται. Τώρα πάμε στα ζανιοκτών. Και ζητώ συγγνώμη για πριν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 44 υπέρ, 27 κατά. Next one. Επόμενη. Στρατηγική προσέγγιση για τα φαρμακευτικά προϊόντα στο περιβάλλον, άρχιτη ψηφοφορία. Πρώτα ψηφίζουμε την προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν. Πέρας της ψηφοφορίας. 70 ψήφοι πέρα. καμία ψήφος κατά και μία αποχή. Τώρα ψηφίζουμε την προφοκέρτηση προς το Συμβούλιο. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. 68 υπέρ, κανείς κατά καμία αποχή. Πάμε στην ψηφοφορία για τη 15η σύμβαση, διάσκεψη συγγνώμη, των συμβαλωμένων μερών, την COP15. Ξεκινάμε με την συμβιβαστική α. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 67 υπέρ, ένας κατά, τρεις αποχές. Εγκρίνεται επομένω. Συμβιβαστική C. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. 66 ψηφί υπέρ. 40, ε, συγγνώμη, 4 κατά και καμία αποχή εγκρίνεται. Προχωρούμε στη συμβαστική Β, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. 63 υπέρ, 4 κατά, 4 αποχές. Εγκρίνεται. Και προχωρούμε. Τροπολογία 34. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. No, it's for show offense, so it's normal that it doesn't work. <laughs> Όχι, είναι λογικό που δεν ε, ανοίγει, λέει ο πρόεδρος, σε σχόλιο μικρόφωνο. 35 τροπολογία, ψήφι υπέρ. κατά. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Άνοιξε τίποτα. Πέρασε. «46 υπέρ, 22 κατά και 3 αποχές». Εγκρίνεται. Προχωρούμε. Συμβαστική B. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική D, ψήφι περ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Z, ψήφι περ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Ψήφι περ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50. Ψήφι περ. Κατά. Να ελέγξουν παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 40 υπέρ, 26 κατά 3 αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 51 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά να ελέγξουμε την 52. πέρας ψηφοφορίας 37 ψήφοι υπέρ 33 ψήφοι κατά μία αποχή εγκρίνεται 53 ψήφοι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική ή e. ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται F. Συμβιβαστική ψήφη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική G. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική S. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 75. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76. Ψήφι υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. So in favor 46 υπέρ, 25 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 77, ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική H, ψήφι περ. κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 81, ψήφι περ. κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική I, J, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J, ψήφι ΠΕΡ, κατά. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Πέρασε ψηφοφορίας. Α, τώρα βλέπετε και εσείς τα αποτελέσματα. 38 υπέρ 19 κατά. Εγκρίνεται. Προχωρούμε. Τροπολογία 97. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 99. Ψήφι περ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική K, K, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. τροπολογία 105, το πρώτο τμήμα μόνο. Εφόσον εγκρίθηκε η συμβαστική D, ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Ε, uh, one. The vote is closed. In favor 42. 42 υπέρ 24 κατά. So we move to 106. 106. Μόνο το πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 46 περί 25 κατά εγκρίνεται. 107 ψήφι περί κατά αποχές εγκρίνεται. 108 περί κατά αποχές εγκρίνεται. 109 περί κατά αποχές εγκρίνεται. 111 μόνο το δεύτερο τμήμα. Ψήφι πέρ. 112 υπέρ. Εκατόν τρία ψήφι υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Ελένα υπέρ. Συμβιβαστική. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Προπολογία 121. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές συγκρίνεται. Συμβιβαστική αίμα. Υπέρ. Κατά αποχές συγκρίνεται. Δεν είναι αυτό. Πώς είναι αυτό εδώ. Συμβαστική όμικρον. ο Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 171-37 προφορική τροπολογία. Να λέει καλή την Ένωση και τα κράτη-μέλη να επαναπροσανατολίσουν τα φορολογικά συστήματα για περισσότερη χρήση της περιβαλλοντικής φορολόγησης. Ποιοι είναι υπέρ αυτής της τροπολογίας προφορικής. Να ελέγξουμε καλύτερα. Άνοιξε, δεν είμαι Είναι αυτό. 42 υπέρ 26 κατά. 138 τώρα ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 139 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική π. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 148. favor, against... Υπέρ. <clears throat> Κατά αποχές εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στην 162. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 163 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 164 υπέρ. Κατά να ελέγξουμε. Αν και νομίζω ότι απορρίφθηκε. Πράγματι απορρίφθηκε. Ταφ συμβιβαστική. Ψήφι υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 170. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. ...171 πρώτο τμήμα, λέει ο πρόεδρος, μόνο. Γιατί έχει εγκριθεί έτσι. Υπέρ κατά. Δεν είμαι βέβαιο για το αποτέλεσμα να ελέγξουμε το πρώτο τμήμα τη 171. Πέρας ψηφοφορία. 54 υπέρ ήταν Συγγνώμη που σας ζήτησα να ελέγξουμε. Προχωρούμε 174 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική γιου. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 179 κατά αποχές εγκρίνεται. We move to compromise Y. In favor, against, abstention. Εκατόν υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 192 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ψήφι περ. Κατά. Να ελέγξουμε το τρίτο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε 35 όλα. Συμβιβαστική W. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική X. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 199. Τροπολογία ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 203. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Okay, so we Έχουμε ψήφιση την τροπολογία Z στην αρχή. Ε, πάμε στη 206. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 207. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική ΑΑ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 211 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική αλφαβήτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στην τροπολογία 216 ψηφίζουμε μόνο το δεύτερο τμήμα Ψήφι Κατά. Να ελέγξουμε. Εγκρίθηκε. 34 προς 29. Πηγαίνουμε στην 217. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1, ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται. 2, ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται. 3, ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται. 4, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, να ελέγξουμε. την 9. Πέραση ψηφοφορίας. 52 υπέρ, συγγνώμη. Τροπολογία 10, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 11, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 12, υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε τη 12. Πέρας. 51 ψήφι πέρ. Αλλά από εδώ δεν ήταν ξεκάθαρο, συγγνώμη. Τροπολογία 13. Ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14. Ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15. Ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 16. Ψήφι πέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 17 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε. Πέραση ψηφοφορίας. 41 ψήφι υπέρ. 18 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 19 ψήφι υπέρ. Κατά. Θέλετε να ελέγξουμε πια τη 18. Ελέγχουμε τη 18. Έτσι έγινε, έτσι ζητήθηκε μάλλον. Απορρίπτεται. Ξαναγυρίζουμε στη 19. Υπέρ της 19 κατά αποχές απορρίπτεται 20 ψήφι υπέρ κατά απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εγκρίνεται συγγνώμη 23. Θέλετε να ελέγξουμε την 22. Αν θέλετε. Ελέγχουμε την 22. Πέραση ψηφοφορίας. Ήταν σαφές. Εγκρίθηκε. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλλά να ελέγξουμε. 24. υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται Ηλεκτρονικά λοιπόν ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. to the next on uh, EU Περνάμε τώρα στην πρωτοβουλία για τους επικονιαστές και ξεκινάμε με την τροπολογία 58. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρα τη ψηφοφορία εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά ίδιοι αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ε, πάμε στην ε, συμβιβαστική 4, ε, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, συμβιβαστική 5, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 86, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην 87 και στην 99 που τις ψηφίζουμε από κενού, ποιοι είναι υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνονται. Συμβιβαστική 6α, υπέρ, κατά. Από... Α, περ κατα 6α, συμβιβαστική 6α. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά, πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά έλεγχος ηλεκτρονικός για την 101. Τέλος. 41 κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά έλεγχος. Α, όχι, συγγνώμη, εγκρίθηκε. 102 τμήμα 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 109. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Έλεγχος για την 109. Τέλος. Απορρίπτεται. 110. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ, 117 επαναλαμβάνει ο πρόεδρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ο, εντάξει, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 117. Πέρας εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 122 υπέρ υπέρ κατά ελέγχουμε ηλεκτρονικός έλεγχος για την 122 What is closed. Rejected. Πέρας απορρίπτεται. Ε, τώρα, η 123 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 126 κατά αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ κατά έλεγχος μάλλον έχει απορριφθεί. Πέρας απορρίπτεται. 128 και 129 είναι ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Καλύτερα να ελέγξουμε, έχετε δίκιο. Ψηφίζουμε, πέρας. Καλά κάναμε και ελέγξαμε. Εγκρίνεται.

κατά «134 και 135». Α, ξαναρχίζω λοιπόν. «134 και 135 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά έλεγχος ηλεκτρονικός». Πέρας απορρίπτεται. Απορρίπτονται μάλλον οι δύο. 136. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Εκρίνεται. 137. 140 μάλλον λέει ο Πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Εκτός και αν θέλετε να ελέγξετε. 142 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 148 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 151 υπέρ κατά έλεγχος απορρίπτεται. Οπότε προχωράμε στην 152 και την 153 ταυτόσημα CPR κατά αποχές εγκρίνονται. Θέλετε να ελέγξουμε, να ελέγξουμε. 152 και 153. Πέρας. Εγκρίνονται. 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 164. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 167. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 166 υπέρ κατά Ας ελέγξουμε 166. Πέρας. Απορρίπτεται. 168. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 169 επέρ κατά αποχές εγκρίνεται 170 επέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός πέρας απορρίπτεται 171 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στις παραθέσεις. Η ένα και οι δύο από κοινού, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 Λοιπόν, 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά ελέγχουμε Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. 27 ελέγχουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά ελέγχος εγκρίνεται τροπολογία 35 υπέρ Κατά. Έλεγχος. Πέρα. Εγκρίνεται. 36 ε, υπέρ. Κατά αποχές ε, ε, ε, εγκρίνεται. Νομίζω. Αλλά αν θέλετε να ελέγξουμε, όχι, εντάξει, εγκρίνεται. 37 Τροπολογία 37. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 38, ε, μάλλον 39, υπέρ, κατά, έλεγχος, γιατί 39, Τέλος, εγκρίνεται. 30, ε, μάλλον, 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά ελέγχουμε 53 πέρας εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική τώρα ψηφοφορία άρχεται Πέρας. Εγκρίνεται. Okay, we move to the next votes on enabling the digital. Πάμε στην επόμενη ψηφοφορία, διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της υγείας και της περιθέψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Συμβιβαστική 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38. Υπέρ. Συγγνώμη υπέρ. Ναι. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά απο... απορρίπτεται. Α, εγκρίνεται. Εγκρίνεται η συμβιβαστική 11. Χρειάζομαι νερό, λέει ο πρόεδρος. 72 υπέρ κατά εγκρίνεται. 73 υπέρ κατά να ελέγξουμε. Πέρες ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάμε στη συμβιβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 81 τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 89 υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. 90 υπέρ κατά αποχή. Να ελέγξουμε την 90. Ελέγχουμε την 90. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 91 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ. Συγγνώμη. 104. Τροπολογία 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην 117. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ συγγνώμη απορρί, αποσύρθηκε 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές κατά αποχές εγκρίνεται 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ένα και δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 και 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 4 και 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 5-9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 6 και 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά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 Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30 υπέρ. 29 συγγνώμη. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά από, να ελέγξουμε 32 πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο του ψηφίσματος άρχεται η ψηφοφορία πέρας Εγκρίνεται. Okay, so the last two votes Οι δύο τελευταίες ψηφοφορίες για το διορθωτικό ψηφοφορία unblock για το πρόστοκο Ριγκέντουμ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συγγνώμη συνάδελφοι, ήταν μεγάλη ψηφοφορία, αλλά πρέπει να πω δύο λόγια για αυτό το διορθωτικό κείμενο, διότι είναι κάπως ασυνήθιστη η κατάσταση. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία. Όπως ξέρετε, τα διορθωτικά κείμενα διορθώνουν τεχνικές πτυχές και συνέχειες αφού ολοκληρωθεί ο τρίλογος. Αλλά αυτή τη φορά Έχουμε... Μας πρότεινε το Συμβούλιο αλλαγές επί της ουσίας του κανονισμού. Ασυνήθιστο. Δεν έχουμε πρόβλημα με την ουσία, διότι οι προτείνομενες αλλαγές σίγουρα θα ε, κλείσουν νομικά κενά. Από την άλλη όμως έχουμε πρόβλημα επί της αρχής, διότι τον αποδεχόμαστε αλλαγές επί της ουσίας του κανονισμού μέσω ενός διορθωτικού κειμένου είναι ε, λάθος ε, στη διαδικασία. Δεν συμβαίνει εντός της καθιερωμένης ε, νομοθετικής διαδικασίας. Οπότε καλήσαμε για ψηφοφορία για να υπάρξει επαρκής πολιτικός έλεγχος από το Κοινοβούλιο, αλλά προτείνουμε να υποστηρίξουμε τα διορθωτικά, διότι έχουμε χρονικούς περιορισμούς. Αυτός ο νέος, αυτοί είναι οι κανόνες που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή μέχρι το Μάιο του χρόνου. Είναι λίγο χαζό που ξεκινήσαμε ε, την νομοθεσία αυτή από το 2012 και ξαφνικά δεν έχουμε χρόνο. Οπότε για να κλείσω, Πρόεδρε, πιστεύω ότι χρήσιμο θα ήταν για εσάς να γράψετε στο Συμβουλίο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζοντας ε, την δυσαρέσκειά μας για τον διαδικασία που ακολουθήθηκε εδώ. Πολύ σαφές, ευχαριστούμε. Ψηφίζουμε το πρώτο διορθωτικό κείμενο ψήφι ΠΕΡ Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερη ψηφοφόρη. Το δεύτερο το διορθωτικό υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και αυτό. Οπότε εδώ ολοκληρώνονται οι ψηφοφορίες για σήμερα. So we start uh, Συνεχίζουμε με το τελευταίο σημείο της μερσιάς διάταξης ε, για σήμερα το πρωί, που είναι στρατηγική προσέγγιση σχετικά με τα φάρμακα στο περιβάλλον. Εκ μέρους του ΕΛΚΑ έχουμε τον κύριο Μπουζόη. Τι προνόμιο να είστε εδώ κύριε Μπουζόη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Φέτο το Μάρτιο έκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανακοίνωσή τη για μια ευρωπαϊκή στρατηγική προσέγγιση σχετικά με τα φάρμακα στο περιβάλλον. Μαζί με του συναδέλφου μου καταρτήσαμε δύο προφορικέ ερωτήσει μία για το Συμβούλιο και μία για την Κομισιόν. Επίση, καταρτήσαμε και ένα ψήφισμα που αν κατάλαβα καλά θα το συζητήσουμε στην Επιτροπή μα τον Ιανουάριο. Η Κομισιόν ορίζει έξι τομεί δράση και αρκετέ ενέργειε συγκεκριμένε. Χρειάζονται περισσότερα όμω σε ορισμένου ε, τομεί ε, πρέπει να επικαιροποιηθεί η νομοθεσία να συμπληρωθεί. Και θα ήθελα μετά τις ερωτήσεις και μετά το ψήφισμά μας θα ήθελα και τα κρατημέλη και η Κομισιόν να αναλάβουν ισχυρέ δεσμεύσει και να προχωρήσουν σε συγκεκριμένε ενέργειε. Νομίζω ότι είναι σαφέ και όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μείωση ε, της ε, επίπτωσης των φαρμάκων στο περιβάλλον, να μειώσουμε τα απόβλητα, αλλά και προληπτικά να εργαστούμε. Όταν αγοράζει ο ασθενή τα φάρμακα, θα μπορούμε να δράσουμε άμεσα. Θα μπορούσε να συνταχογραφούνται τα φάρμακα με βελτιστοποιημένη συσκευασία, λαμβάνοντα υπόψη τις ανάγκες. Θα μπορούσαμε να βρούμε πολλές λύσεις για νοσοκομεία, για φαρμακεία, αλλά κατ' εμέ αυτό που χρειάζεται είναι μεγαλύτερη δέσμευση και προσήλωση στη μείωση της επίπτωσης των φάρμακων στο περιβάλλον. Αυτά και περιμένω να ακούσω σήμερα τη συζήτηση και κυρίως να ακούσω τις απαντήσεις που θα μας δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ο κύριος Ζίντελ. Νομίζω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες αναγνωρίζουν ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα και να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις ε, για τα φάρμακα στο περιβάλλον. Και αυτό είναι θετικό. Έχουμε το πρόβλημα της ε, μικροβιακής αντοχής ε, και ε, στην ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου βλέπουμε ότι χιλιάδες άνθρωποι είχαν τη ζωή τους από λοιμώξεις λόγω των ε, βακτηρίων ε, που ανθίστανται στα αντιβιωτικά. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και ένα άλλο πρόβλημα είναι οι εκπομπές και η έκθεση των υπόγειων και επίγειων υδάτων σε αυτές τις φαρμακευτικές ουσίες. Είναι θετικό που όλες οι πολιτικές ομάδες θέλουν ε, να πετύχουμε κάτι ε, σε αυτά τα θέματα, με αυτό με δράσεις ε, και της ενέργειας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και μέσω του δικού μας ψηφίσματος. Ευχαριστώ. Λενουάρ για την Κομισιό. Για, την, για το Ρινιού. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να συζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι ανάγκη να υπάρξουν προληπτικά μέτρα για κάποια επικίνδυνα φάρμακα, για τα, τα αντικαρκυνικά για παράδειγμα, ε, χορηγούνται από στόματος αυτή τη στιγμή, που σημαίνει ότι για την απαλήφη τους, ε, τη διάθεσή τους, ε, έχουμε προβλήματα. Ρήπανση του περιβάλλοντος, ε, και γενικότερα μπορεί να προκύψουν και άλλοι καρκίνοι μακροπρόθεσμα λόγω της μη σωστής διάθεσης αυτών το φαρμάκο. Ευχαριστώ. ID. Δεν βλέπω κάποιον. Μισελ Ριβασία, eh Ακούστε. Δεν ξέρω αν είναι αργά για να πάρουμε μέτρα. Ήδη από το 2008 το έχουμε θέσει το θέμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από τότε είχε πει ότι πράγματι έχουμε θέμα με τα φάρμακα στο περιβάλλον και κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Μετά, το 2013, κυκλοφόρησε μια μελέτη που λέει ότι πρέπει να ληφθούν μαθητικά μέτρα και η Επιτροπή θα καταθέσει προτάσεις μέχρι το 2015. Σήμερα έχουμε 2019. Τι μας προτείνει η Κομισιόν ε, μια extra light στρατηγική. Πάρα πολλά τα κίνητρα να κινήσουμε, θα ήταν καλό να ενημερώσουμε κτλ. κτλ. Σας ενημερώνω ότι ο ΣΑ σε έκθεση του λέει πρέπει να ληφθούν δρακόντια μέτρα και μέτρα νομοθετικού περιεχομένου. Άρα τι light. Δεν χρειαζόμαστε κάτι light εδώ. 10% των φαρμάκων μπορεί να βλάπτει το περιβάλλον, λέει έκθεση ορμόνες, αντικαταθλιπτικά, αναλγητικά φάρμακα είναι τα χειρότερα. Υπάρχει υπερσυγκέντρωση στα λίματα που μπορεί να δημιουργήσει μικροοργανισμούς, ανθεκτικούς στα φάρμακα και μάλιστα είναι ένα θέμα που ετέθη υπόψη της ομάδος των 20, των G20 και πρέπει να ληφθούν μέτρα κατεπήγοντα. Άρα, τρία πράγματα θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Πρώτο πώς επηρεάζουν το περιβάλλον τα φάρμακα σε επίπεδο αδειοδότησης, έγκριση κυκλοφορίας. Όταν ένα φάρμακο παίρνει άδεια, θα πρέπει να βλέπουμε τι κινδύνους ενέχει αυτό για το περιβάλλον. Όπω ήδη συμβαίνει για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Δεν συμβαίνει όμω αυτό για τα φάρμακα που προορίζονται για χρήση από τον άνθρωπο. Αυτή θα ήταν μια πρόταση πολύ σημαντική και όχι θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν, πρέπει να συμπεριληφθούν. Δεν είμαστε στην ευκτική τώρα. Είναι light αυτό. Πάμε στο δεύτερο. Πρέπει, γιατί σε όλα τα φάρμακα ε, υπάρχουν 3.000 περίπου δραστικές ουσίες που θα πρέπει να τις ε, εξετάσουμε. Υπάρχει αξιολόγηση κινδύνου για ό,τι φάρμακο κυκλοφόρησε μετά το 2006, όχι όμως για τι γίνεται πριν το 2006. Χρειάζεται όμως αυτό. Επίσης, η Κομισιόν πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η παρασκευή εισαγόμενων φαρμάκων να ανταποκρίνεται στα ίδια υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν για την παρασκευή φαρμάκων εντός Ένωσης. Γιατί με την ιστορία αυτή της αγωγής ε, δραστικών νησιών βλέπουμε ότι κυρίως στην Ινδία και στην Κίνα παρασκευάζονται. Άρα εδώ έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εμείς ζητάμε τρακόντια μέτρα για το περιβάλλον, πολύ καλό αυτό, αλλά τι γίνεται με εκείνες τις χώρες, άντε γεια. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν μέτρα και ναι με να εγκρίνεται η εισαγωγή τέτοιων φαρμάκων, αλλά να υπάρχει έλεγχος και έγκριση. Γιατί δεν είναι καλό για τις χώρες αυτές, ούτε και για μας. γιατί και στα τρόφιμα και στο περιβάλλον ε, βρίσκουμε από, μολυσμένα, ε, από τα μολυσμένα νερά ε, υπολείμματα αυτών των φαρμάκων. Θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Αλλά πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί σε αυτά που ζητάμε, γιατί αλλιώς δεν θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ιωάννα Κουτσίνσκα, για το ΣΥΑΡ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ πολύ πολύ θετικό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται για την παρουσία, την ύπαρξη των φαρμακευτικών δραστικών ουσιών στο περιβάλλον. Είναι εξαιρετικά θετικό. Το κείμενο είναι ιδιαίτερα κέριο, πολύ καλά συντεταγμένο. Ευχαριστώ τη Γραμματεία και τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν μαζί μας. Υποστηρίζω τις ε, περισσότερες ε, τροπολογίες, ιδιαίτερα αυτούς που αυτές που αφορούν την παραγωγή λιγότερων νοσηρών φαρμάκων. Ε, θα πρέπει να προωθήσουμε μια νέα συνείδηση για την παραγωγή, αλλά και για μετά την παραγωγή μέσω νέων πρακτικών που ρυθμίζουν λιγότερο το πλαίσιο παραγωγής, αλλά περισσότερο συγκεντρώνονται στα σε επιπτώσει των φαρμάκων αυτών όταν αυτά έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον. Νέο είδου ευαισθησία, νέο είδου συνειδητοποίηση της σημασία της νοσηρότητα των δραστικών ουσιών των φαρμάκων στο περιβάλλον. Ω Ευρωκοινοβούλιο οφείλουμε να στηρίξουμε τους ε, φορείς που είναι δεσμευμένοι στην προστασία του περιβάλλοντος και όλα αυτά σεβόμενοι βέβαια την ε, ελευθερία πρόσβασης των ε, ασθενών στα φάρμακα και χωρίς να αποδυναμώνεται η έρευνα. Μάλιστα αυτό το αναφέρουμε στο 21-27 του ψηφίσματος. Με άλλα λόγια θα πρέπει να ενεργήσουμε για να μειωθεί ο κίνδυνος που προκαλείται από την παρουσία των φαρμάκων στο περιβάλλον, σεβόμενη όμως την πρόσβαση στα φάρμακα των ασθενών. Αυτό το οποίο ε, λείπει κατά τη γνώμη μου από αυτό το ψήφισμα είναι ότι δεν γίνεται λόγος για την φαρμακευτική βιομηχανία, διότι είναι αυτή που θα πρέπει να αναγνωρίσει τα προβλήματα της ελλείψης τόσο για τα ε, φάρμακα για τα ζώα όσο και για τα ε, φάρμακα προς ανθρώπινη κατανάλωση. Μιλώ ας πούμε για ε, τις αντιδράσεις που γίνονται μέσω αυτών των δραστικών ζώων που πολλές φορές συνεχίζονται για πολλά χρόνια και μέσα στο νερό και μέσα στη γη. Σας ευχαριστώ και θα υποβάλω σχετικές τροπολογίε. Ευχαριστώ. Εξ ονόματο της ΚΟΕ δεν υπάρχει ομιλητής. Όχι. Υπάρχει κάποιο άλλος που θα θέλει να πάρει το λόγο πριν να δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Και πάλι όχι. Ωραία λοιπόν, οπότε ε, το λόγο έχει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ή εκπρόσωπος της Επιτροπής, κυρία Ντεζέρ. Σας ευχαριστώ πολύ. Από την ε, πλευρά της Επιτροπής καταρχώς θέλω να πω ότι είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που το Ευρωκοινοβούλιο έχει ενδιαφερθεί τόσο πολύ για το θέμα των φαρμάκων. Όπως γνωρίζετε, η νέα Επιτροπή ανέλαβε καθήκοντα μόλις αυτή τη Δευτέρα και ο η, νέος, η νέα πρόεδρος, η κυρία Βοντερ Λάγεν, έχει δώσει κατευθυντήριες γραμμές πολιτικού τύπου. Ήδη πριν από λίγο καιρό έχει ανακοινώσει το πράσινο σύμφωνο, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και τη φιλοδοξία για μηδενική ρήπαση. Πιστεύουμε ότι το θέμα των φαρμακευτικών προϊόντων θα μας απασχολήσει πολύ, γιατί έχουμε αυτό το νέο πλαίσιο και είναι πραγματικά σπουδαίο που όλοι σας ενδιαφέρεστε και ε, θέλετε να συνεργαστούμε. Επίσης είμαστε ευτυχείς γιατί πολλά από τα θέματα που αναφέρονται στο σχέδιο ψηφίσματος ε, στην ουσία αντικατοπτρίζουν αυτό που περιλαμβάνεται στη στρατηγική μας για τα φάρμακα. Όπως γνωρίζετε αυτή η στρατηγική εγκρίθηκε το Μάρτιο από την Επιτροπή και έκτοτε έχουμε αρχίσει δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ προέρχομαι από την DG Περιβάλλον αλλά συνεργάζομαι με τους ε, ε, συναδέλφους από την DG Υγεία, Υγεία και Καταναλωτές. Θέλουμε να δουλέψουμε για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των φαρμακευτικών προϊόντων και αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο από την πλευρά του περιβάλλοντος. Εγώ είμαι υπεύθυνη για το νερό και από τη στιγμή που αυτές οι ουσίες έχουν μπει ήδη στο νερό είναι πολύ δύσκολο να τις αφαιρέσουμε. Γι' αυτό πρέπει να αρχίζουμε δουλειά πολύ νωρίτερα ώστε να εξασφαλίσουμε πως δεν θα φτάσουν στο νερό. Ε, τούτου λεχθέντος, ε, μία από τις βασικές αρχές ε, πίσω από τη φαρμακευτική μας στρατηγική είναι βεβαίως ότι εκείνοι που χρειάζονται ειδική θεραπεία, ειδική και οι φαρμακευτικοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτήν. Η Κομισιόν λοιπόν δεν θέλει με κανένα τρόπο να περιορίσει τη δυνατότητα κυκλοφορίας αυτών των φαρμάκων που χρειάζονται, ειδικά για πολύ ε, σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος που αναφέρθηκε εδώ. Όλα αυτά λοιπόν αναφέρονται σε διάφορους ε, τομείς, ε, Αναφέρουμε και διάφορους τομείς όπου πρέπει να υπάρξει δράση κατά τη γνώμη μας και αναζητούμε τρόπους βιώσιμους για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δραστικές ουσίες. Έχουμε αρχίσει ενέργειες σε διάφορους τομείς, όπως αναφέρθηκε όταν ε, ε, ο Επίτροπος θα χρειαστεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα θέματα, θα δώσουμε όλες τις λεπτομέρειες και την κατάσταση πρόοδου. Θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να σας ενημερώσω ότι ε, διοργανώνεται στη Σαραγώσα μια μεγάλη διάσκεψη για το νερό και είναι αφιερωμένη στα φάρμακα στις 12 Δεκεμβρίου μία συνεδρίαση και θα συζητήσουμε με εκπροσώπους της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Ελπίζω πως τουλάχιστον κάποιοι από εσά θα μπορέσετε να συμμετέχετε σε αυτή τη διάσκεψη. Θα μεταδίδετε τη διασκεψη θα αναμεταδιδετε απευθειας και στο διαδίκτυο, οπότε θα μπορούσατε ίσως να το παρακολουθήσετε μέσω του διαδικτύου. Λίγες περισσότερες λεπτομέρειες τώρα για κάποια από τα ζητήματα που αναφέρθηκαν. το ένα αφορούσε το περιβαλλοντικό αντίκτυπο και την αξιολογή, τις αξιολογήσεις που γίνονται και ίσως τις διαφορετικές προσεγγίσεις ε, όσον αφορά τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση και τα φάρμακα για τα ζώα, για τα φάρμακα για τους ανθρώπους θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως οι ασθενείς θα έχουν την καλύτερη δυνατή αγωγή και ε, προσιτή. Η διαφορετική προσέγγιση δεν σημαίνει πως δεν εκτιμούμε και δεν αξιολογούμε την περιβαλλοντική, ε, τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των ανθρωπίνων φαρμάκων. Εδώ εστιάζουμε περισσότερο στο τομέα της αντιμετώπισης, ε, της άβλησης των μάλλον της μετρίασης των επιπτώσεων. Ε, στη, κάθε εταιρεία κάνει μια τέτοια εκτίμηση για κάθε φάρμακο το οποίο προτείνει. Επίσης ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και να κατανοήσουμε ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα χημικά δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο στο πλαίσιο της, ε, του ευρωπαϊκού νομικού οπλοστασίου. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας όταν μιλάμε για φάρμακα. Ε, Επίση, αναφέρθηκε πως η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει νομοθετική δράση. βεβαίω. δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά σύμφωνα με την, μάλλον με τη βάση την νομοθεσία περί υδάτων έχουμε ρυθμίσει κάποια θέματα για τα φάρμακα. Ας πούμε έχουμε την οδηγία περί παραβολοντικών ε, προδιαγραφών και εδώ ήδη αναγράφονται τα φάρμακα στον αποκαλούμενο κατάλογο παρακολούθησης όπως λέγεται. Ε, ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε δύο και στην επόμενη ενημέρωση ελπίζω πως θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες φαρμακευτικές δραστικές ουσίες όπως κατανοείτε όμως πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία συμμετέχουν τα κράτη-μέλη και εσείς και ελπίζουμε πως θα είμαστε σε θέση όταν θα έχουμε ενημερωμένο κατάλογο των ουσιών προτεραιότητες μέσα στην προβλεπόμενη διαδικασία μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την κατάλληλη στιγμή και να εξασφαλίσουμε ότι θα ε, έχουμε περισσότερες ουσίες στον κατάλογο παρακολούθησης. Επίσης, σε διεθνές επίπεδο υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει. Συνάδελφοι από την DG Υγεία ε, βρίσκονται σε επαφή με κάποιους από τους κύριους εταίρους σε αυτά τα ζητήματα. Και από την πλευρά μας, από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος κάνουμε το ίδιο. Νομίζουμε πως είναι πολύ σημαντικό να το συζητήσουμε όχι μόνο με τις αρχές αλλά και με την βιομηχανία, τη φαρμακοβιομηχανία. Ε, και να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα πιέσουμε και τους φαρμακοβιομήχανους ε, ένα από τους καλύτερους τρόπους ήταν, ε, είναι, πιστεύουμε, η ε, πράσινη διαγωνισμοί. σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και για το ενδιαφέρον σας. Ευχαριστούμε. Το επόμενο βήμα θα είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 29 Ιανουαρίου. Ο κύριος Μπέζερ μπορεί να μην είναι μαζί μας τότε. Θα παραμένετε αναπληρωματικό μέλος ε, της... Α, ωραία. Ωραία, εδώ κλείνει το πρωινό τμήμα της συνεδρίασης. Θα συνεχίσουμε στις 2 και 40.